Επίσης, για την Δευτέρα το βράδυ, για την Δευτέρα το απόγευμα. Όχι. Τρίτη. Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, οι έξι εκθέσεις κωδικοποίησης Ντούντα που προβλέπεται να ψηφιστούν την Τρίτη θα ψηφιστούν σε μια μεταγενέστερη σύνοδο ολομέλειας. Υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά. Συμφωνείτε οι εκθέσεις Ντούντα να μεταφερθούν σε μια μεταγενέστερη ολομέλεια. Εντάξει. Από πολλές ομάδες έχω λάβει μια αίτηση για συζητήσεις για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν με ψήφισμα, με καταληκτικό ψήφισμα. Τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ τους πολιτικές ομάδες ποιος θα λάβει το λόγο, γιατί όλοι οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο, θέλουν να το παρουσιάσουν συγχρόνως. Κύριε Λάμπερτς, φαντάζομαι ότι και εσείς θέλατε να λάβετε το λόγο. Ο κύριος Πιτέρα και η κυρία Τσίμερ επίσης μπορούν να λάβουν το λόγο υπέρ, αν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο κατά και μετά θα ψηφίσουμε. Κύριε Πιτέλα, παρακαλώ, υπέρ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρο. Όπως ε, προείπατε, προβλέψατε, η ομάδα μας είναι υπέρ του να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας του Ιανουαρίου το ψήφισμα που κλείνει τη συζήτηση για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Γιατί είναι σωστό το Κοινοβούλιο να πει τη γνώμη του, να επιβεβαιώσει τις προτεραιότητες του και εμείς ως ε, σοσιαλιστές δημοκράτες να μπορέσουμε να υποδείξουμε τις προτεραιότητές μας που είναι το περιβάλλον και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Ευχαριστώ. Κύριε Λάμπερτς, για το θέμα. Όχι, κύριε Πρόεδρε, μπορεί σε κανέναν να αρέσει πολύ το θέατρο, αλλά χρειάζεται το Κοινοβούλιο να εκφραστεί μέσω ψήφου για το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η πιο σημαντική τη πράξη. Άκουσα στη διάσκεψη του Πρόεδρου να λένε κάποιοι, να εντάξει, θα λάβουμε θέση για το πρόγραμμα του 2015. Δηλαδή, εκλογέ, ευρωεκλογέ, νέα επιτροπή, και το κοινοβούλιο μα 18 μήνε αργότερα θα πει τη γνώμη του. Είναι γελίο κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι το αργότερο τον Ιανουάριο πρέπει να ψηφίσουμε για ένα ψήφισμα ε, όσον αφορά το πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν, εάν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει αυτό εδώ το θεσμικό όργανο. Καλώ. Ο κύριο Πιτέλα ζήτησε να γίνει αυτό τον Ιανουάριο. Ποιο υποστηρίζει την πρόταση του κυρίου Πιτέλα. Υπέρ, υπέρ. Κυρία Τσίμερ, και εσείς υποστηρίζετε την πρόταση του κυρίου Πιτέλα ή θέλετε να γίνει το Δεκέμβριο η ψηφοφορία αυτή. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης Πιτέλα για τον Ιανουάριο. Φερχόστα. κύριε, Πρόεδρε. Πρόεδρε, τον Ιανουάριο θα ήταν σωστό για να μπορεί να γίνει η συζήτηση αύριο και να προετοιμάσουμε το ψήφισμα καταλήλως. Αλλά ζητάω μόνο να μην είναι φάρσα ή χριστουγεννιάτικο δέντρο παραφορτωμένο. Ξέρω ότι ε, αυτό φοβάμαι εγώ τουλάχιστον. Να είναι 10 σελίδες, 15 σελίδες, 20 σελίδες με όλες τις προτεραιότητες. Όχι. Να είναι ένα σύντομο πολιτικό ψήφισμα. Τότε υποστηρίζω την πρόταση του κυρίου Πιτέλα. Θέλετε, κύριε Ζάε, να μιλήσετε ενάντια στην πρόταση Πιτέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προτιμούσα να διατηρήσω τη λογική διαδικασία ένας ομιλή υπέρ, ένας ομιλή κατά και μετά ψηφίζουμε. Το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, ιδίως τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και το έχει μόνο η Κομισιόν. Η χρονιά όμως η φετινή είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και δεν προβλέπει το πρόγραμμά μας ένα ψήφισμα γιατί η Κομισιόν ανέλαβε το έργο της μόνο την 1η Νοεμβρίου. Δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία ενός ψηφίσματος το Σεπτέμβριο και μετά ε, να αναλάβει η Κομισιόν και να συνεχίσει εγώ νομίζω ότι μετά από ένα έτος εκλογών αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι πραγματική εργασία. Όχι ψηφίσματα, όχι ψηφίσματα για ένα πρόγραμμα το οποίο θα εγκρίνει αύριο η Κομισιόν. Η δική μου πρόταση λοιπόν είναι να μην υπάρξει ψήφισμα και να ξεκινήσουμε την εργασία μας. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά αγαπητέ συνάδελφε, βάσει της ε, ημερήσια διάταξης βάσει του κανονισμού μάλλον πρέπει να ακολουθήσουμε μια σωστή διαδικασία. Υπάρχει μια πρόταση του κυρίου ε, Πιτέλα και έχουμε και την πρόταση της κυρίας Τσίμερ η οποία θέλει να υπάρξει το ψήφισμα και συζήτηση αυτή τη βδομάδα. Πρέπει να δώσω λοιπόν το λόγο σε αυτούς οι οποίοι θέτουν τις προτάσεις αυτές. Η κυρία Τσίμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Για να είμαι και, εμεί, και εγώ σαφής. Η δική μου πολιτική ομάδα έχει ζητήσει και στο παρελθόν η δήλωση αυτή η οποία θα γίνει αύριο από την Κομισιόν να ακολουθηθεί από ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους εξής λόγους. Πρώτον, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο έτος της Κομισιόν. Δεύτερον, όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν δώσει γνωμοδοτήσεις σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της δράσης της Κομισιόν και το πρόγραμμα εργασίας το 2015. Και τρίτον, στην συνέλευση των Προέδρων έχει γίνει μια συζήτηση με τον κύριο Γιούνκερ, με τον κύριο Τίμερμαν και οι πολιτικέ ομάδε έχουν λάβει ήδη υπόψη πώ θέλει η Κομισιόν να προχωρήσει για τα θέματα αυτά και επίση η Κομισιόν έχει το λεγόμενο, τον διαβόητο killing list, τον κατάλογο των προτάσεων που δεν θα ευδοκιμήσουν και υπάρχουν πολλές ε, διαμαρτυρίες από το Κοινοβούλιο ότι προγράμματα όπως αυτά για, την, ε, για το, ποιότητα της ατμόσφαιρας του αέρα δεν θα πρέπει να αφαιθούν να μείνουν χωρίς πρόθεση από την Κομισιόν. Ποιος είναι υπέρ της προτάσεως της κυρίας Τσίμερ, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Όχι. Πριν. Πριν κάνουμε την ψηφοφορία. Αγαπητές συνάδελφες, πρέπει να υπάρχει κάποιο ο οποίο να ψηφίσει υπέρ, να ομιλήσει υπέρ τη πρόταση τη κυρία Τσίμερ και να ομιλήσει κάποιο άλλο κατά. Υπέρ. Ο κύριο Λαμπέρ. Αν θέλουμε να έχουμε τον οποιοδήποτε αντίκτυπο σε αυτά που θέλει να κάνει η Κομισιόν, όσο το ταχύτερα τόσο και καλύτερα. Αν λοιπόν ήδη από το Δεκέμβριο να ψηφίσουμε, α το κάνουμε τώρα. Αν δεν το κάνουμε το Δεκέμβριο, το κάνουμε τον Ιανουάριο. Αλλά αν υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ του Δεκεμβρίου, α το κάνουμε τώρα. Κατά. Ποιο θέλει να λάβει το λόγο κατά αυτή τη πρόταση. Ωραία. Οπότε έχουμε την απότατη πρόταση η οποία είναι να ψηφίσουμε τώρα, αυτή τη βδομάδα. Είναι η πρόταση της κυρίας Τσίμερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η πρόταση αυτή. Η πρόταση του κυρίου Πιτέλα για τον Ιανουάριο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γίνεται δεκτή η πρόταση. Εντάξει, να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Όχι. Πέρας ψηφοφορίας. ...231 υπέρ, 121 κατά, 18 εποχές. Τετάρτη. Οι πράσινοι ζητήσανε να υπάρξει μια δήλωση της ΥΠΑ, του, ΥΠΑ εκπροσώπους σε σχέση με την, ε, τις πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία, όπως ανέφερα προηγουμένως. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Χάμς, η οποία έχει καταθέσει αυτή την πρόταση από τους πράσινους. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήδη έχετε κάνει αναφορά στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι όλοι μας όταν ακούσαμε για αυτή την ενέργεια στην Τουρκία πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί και εκπλαγήκαμε για αυτές τις επιθέσεις κατά του τύπου της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Πρέπει να ξέρουμε ότι ήδη υπάρχει μια αντική πορεία σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και πριν από τα, πρόσφατα γεγονότα, ακόμα και πριν από το Γκεζί Πάρκ, γιατί τότε είχαν ρηχτεί στη φυλακή αντιφρονούντες δημοσιογράφοι γιατί είχαν άποψη κατά τη κυβέρνηση. Η περίπτωση του Γκέζι Πάρκ μα έδειξε πραγματικά την υπαναχώρηση που έχει γίνει σε σχέση με τα δικαιώματα του τύπου στην Τουρκία. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και γι' αυτό θεωρώ ότι η πρόταση των άλλων ε, πολιτικών ομάδων να υπάρξει ένα ψήφισμα μόνο τον Ιανουάριο, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Ο κύριος Λεγιαρίκ από την ΚΟΕ. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε στην αρχή της συνεδρίας, ίσως αφορά την ελευθεροτυπία στην Τουρκία. Πιστεύω πως πρόκειται για μια ενέργεια εξαιρετικά σημαντική και ισχυρή, στεναρή. Τα όσα έγιναν εχθές στην Τουρκία είναι πραγματικά παράδεκτα, γιατί σε 13 πόλεις από ό,τι φαίνεται συλλήφθηκαν ε, δημοσιογράφοι και ε, κυκλοφορούν ε, απειλές μέχρι τα Χριστούγεννα. Για 150 δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων οι κύριοι δημοσιογράφοι του, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και των πιο μεγάλων εφημερίδων. Παρακαλώ λοιπόν να γίνει η παρέμβαση της ΥΠΑ της εκπροσώπου ή κάτι εν για να σταματήσει αυτή η κατάσταση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ υπάρχουν ε, θέσει εναντίον. Ο κύριο Λάμστορφ. Δεν θα μιλήσω κατά. Εγώ θέλω να μιλήσω υπέρ της πρότασης της κυρίας Χάμς. Αλλά αυτό το οποίο λέει ο κύριος ε, Ιαρίκ να ψηφίσουμε ήδη με ένα ψήφισμα αυτή τη βδομάδα Νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό που πρότεινε η κυρία Χάμ, Αυτή τη βδομάδα συζήτηση και τον Ιανουάριο ένα ψήφισμα. Και αυτό δεν ήταν ακριβώ ε, αυτό που έπρεπε να γίνει ο κύριο Μέσερσμιτ, γιατί πρέπει να μιλήσει κάποιο εναντίον. Υποθέτω ότι θα μιλήσετε εναντίον, κύριε Σμιτ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι κατά της πρότασης της κυρίας Χάμς ή όχι. Κατά. Το σπλίτ θα το κάνουμε μετά, την διαφοροποίηση. Θέλει να μιλήσει κανείς κατά, εάν όχι, εντάξει. Λοιπόν, <clears throat> ας ψηφίσουμε για την συμπερίληψη αυτού του σημείου στη μέση διάταξη. Ποιο είναι υπέρ τη συμπερίληψης. Κατά. Αποχές. Γίνεται δεκτό να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στη μέση διάταξη. Τώρα το ερώτημα είναι πότε ποιοι θέλουν η συζήτηση αυτή με ψήφισμα να γίνει με ψήφισμα. Ψήφι υπέρ. Ξαναλέω έχουμε αποφασίσει να γίνει συζήτηση και πρέπει να δώσει την άποψή τη. η ύπατη εκπρόσωπος. Το επόμενο ερώτημα είναι αν θα πρέπει η συζήτηση αυτή να ακολουθηθεί από ψήφισμα. Ποιος θέλει ένα ψήφισμα στο τέλος τη συζήτηση. Κατά. Αν δεν γίνει αυτή τη βδομάδα, πότε θα γίνει αυτό, λέει ο πρόεδρος. Ωραία πάρα πολύ συγκεκριμένα. Κυρία Χάλς, ζητήσατε για αυτή τη βδομάδα ή για τον Ιανουάριο. Εγώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει την άποψή του το ταχύτερο δυνατό. Αλλά με ενδιαφέρει να είναι και αποφασιστική η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε τακτικό επίπεδο αυτή τη εβδομάδα και να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αυτό ήταν αυτό το οποίο καταλάβαμε από αυτά που είπατε. Λοιπόν, επομένω, εάν συμφωνούμε όλοι, αυτή τη βδομάδα θα γίνει συζήτηση και τον Ιανουάριο θα εκδώσουμε ένα ψήφισμα. Λοιπόν, να ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Ποιο είναι υπέρ του να γίνει το ψήφισμα τον Ιανουάριο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία, είναι σαφές επομένως. Το ψήφισμα θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο. Η ομάδα του ECR, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, θέλουν να υπάρξει την πέμπτη, για την πέμπτη αναβολή του ψηφίσματος για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ο κύριος μέσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν πως πρόκειται για πολύ λεπτό θέμα και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να διαπραγματευτούμε τις συμβιβαστικές του για το ψήφισμα. Εξ ονόματος του ECR θα ήθελα να προτείνω να παραταθεί η προθεσμία μέχρι τις, ε, την, την Τετάρτη στις 11 η ώρα, ώστε να ψηφίσουμε αυτή τη βδομάδα, αλλά την Πέμπτη. Ποιο υποστηρίζει την πρόταση του κυρίου Messerschmidt υπέρ τη πρόταση κανεί. Θέλει κανείς να μιλήσει κατά της πρότασης του κύριου Μέσιο Σμιτ. Παρακαλώ, κύριε Άντες. Ήδη καθυστερήσαμε υπερβολικά από τον περασμένο μήνα σε αυτό το μήνα και είχαμε πάρα πολύ χρόνο για να συμφωνήσουμε σε ένα ψήφισμα κοινό και γι' αυτό είναι σωστό να μείνουμε στο χρονοδιάγραμμά μας έχουμε δουλέψει με βάση αυτό και απορρίπτουμε απόλυτα το, η πρόταση να ψηφίσουμε την Πέμπτη πρέπει να το ψηφίσουμε την Τετάρτη όπως ε, είναι στην ημερήσια διάταξη Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα την πρόταση του κυρίου Μέσοσπιτ αναβολή της ψηφοφορίας την Πέμπτη. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης του κυρίου Μέσοσπιτ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η πρόταση του κυρίου Μέσοσπιτ. Οπότε έχουμε καθορίσει την ημέρα για διάταξη της εβδομάδα αυτής, λέει ο πρόεδρος. και ερχόμαστε στην, σύμβαση, στην σύσταση της κυρίας Αγιούσο για τη συμφωνία σε σχέση με το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Η κυρία Έστερ Χεράνς θα αντικαταστήσει